So, guten Morgen, Καλημέρα συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε. Έχουμε ένα έργο μαμούθ μπροστά μας. Ψηφοφορία για ε, τα οπτικοακουστικά μέσα και την ε, αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας. Θέλω όμως να ξεκινήσω με τα βασικά τα διαδικαστικά. Περνάμε στο πρώτο ε, θέμα της ημερήσιας διάταξης, έγκριση αυτής. Εγκρίνεται η σε διάταξη. Υπάρχουν αντιρρήσεις, ενστάσεις. Είναι οφθαλμοφανές πως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Εγκρίνεται λοιπόν. Θέμα 2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 23ης και 24ης Ιανουαρίου 2015. Το σχέδιο των πρακτικών το έχετε λάβει στα έγγραφά σας κάπου εκεί κρυμμένο μέσα στη, στα έγγραφά σας είναι. Προτείνω τα πρακτικά να θεωρηθούν εγκεκριμένα εφόσον μέχρι το τέλος της συνεδρίασής μας σήμερα δεν υποβληθούν ενστάσεις και αντιρρήσεις. Ελπίζω να συμφωνείτε. Τρία. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Πρώτον, έχουμε διερμηνία στη διάθεσή μας για τις εξής γλώσσες. Γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, εσθονικά, ουγγρικά, πολωνικά, σλοβενικά, βουλγαρικά και ρουμανικά. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο σήμερα, όπως πάντοτε. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι οι αποφάσεις των συντονιστών της 22ης Μαρτίου που σας απεστάλησαν στις 24 Μαρτίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί αν έως, ε, μάλλον όχι, ε, επρόκειτο να θεωρηθούν εγκεκριμένα αν έως τις 28 Μαρτίου δεν είχαν υποβληθεί αντιρρήσεις. Αυτό δεν συνέβη, επομένως θεωρούνται εγκεκριμένες οι αποφάσεις των συντονιστών. Προτού περάσουμε στην ε, ψηφοφορία, ο κύριος Γραμματικάκης ζήτησε να του δώσω το λόγο σύντομα, προκειμένου να μας ενημερώσει σχετικά με μια πολύ όμορφη και πολύ ενδιαφέρουσα ε, εκδήλωση. Γιώργο, πολύ γρήγορα όμως. Έχεις το λόγο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, είπατε πολύ όμορφη και πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Πράγματι, πληροφορώ όλους τους συναδέλφους ότι στις 3 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, υπάρχει ολόκληρη την ημέρα μια εκδήλωση που ονομάζουμε «Τριλογία ελληνικού πολιτισμού». Μια ομιλία στις 12.30 από ένα διακεκριμένο καθηγητή σχετικά με την Ευρώπη και την επίδραση των αρχαίων ε, ελληνικών ε, γραμματείας στη σύγχρονη Ευρώπη. Δεύτερο, μια έκθεση φωτογραφίας από ελληνικά νησιά και τρίτο το βράδυ στις 7 η ώρα μια παράσταση της εθνικής λυρικής σκηνής σε μουσική του Μοντεβέρντι. Νομίζω ότι όλοι θα ευχαριστηθείτε την ημέρα και θα χαρώ να σας δω όλους εκεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την ενημέρωση και κυρίως για την διοργάνωση αυτής της εξαιρετικής εκδήλωσης την οποία και θα έχουμε την ευκαιρία να απαλλάψουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Περνάμε αμέσως στην ψηφοφορία. Βλέπετε μπροστά σας αυτόν τον ε, χοντρό πάκο που έχετε μπροστά σας και τον κατάλογο ψηφοφορίας. Το σχέδιο ε, έκθεσης για την ε, οδηγία για τα οπτικοακουστικά παρουσιάστηκε από τις δύο συνεισηγήτριες 19 Οκτωβρίου 2016 ήταν η προθεσμία υποβολής ε, των τροπολογιών. 950 προήλθαν από την δική μας Επιτροπή και μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών Ένβιο, Ίμκο, ΛΥΜΠΕ και Γιούρι έχουμε ένα σύνολο σχεδόν 1400 τροπολογιών, κάτι που υπογραμμίζει και το μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την νομοθετική πρόταση. Χωρίς το εξαιρετικό έργο και την υποστήριξη του Στέφανη Μπιαζόλη και της Φραντσέσκα Μπιαζόλη, όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά και θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ε, ιδίως την Στεφανή για το υπεράνθρωπο έργο της και την προσπάθεια που κατέβαλε για, αυτό το εξαιρετικό, για αυτή την εξαιρετική δουλειά. Την ευχαριστούμε και εκείνοι και όλους τους άλλους που εργάστηκαν επί του θέματος αυτού θερμότατα. Να ευχαριστήσω επίσης φυσικά και όλους τους σκιώδεις και τους βοηθούς αλλά και τους δικούς μας ε, ε βοηθούς Κατερίνα Μάγκολ και Τίνο Κούναρτ οι οποίοι επίσης εργάστηκαν σκληρότατα. Είχαμε πολύ έντονες ε, συζητήσεις και στη συνεδριάση των σκιωδών, αλλά νομίζω ότι στο τέλος της διαδικασίας καταφέραμε να καταλήξουμε σε πολύ καλούς συμβιβασμούς. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στη Ζαμπίνη Φερχάιν τώρα και μετά να περάσουμε στη ψηφοφορία. Ζαμπίν, Ναι, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμματεία, ιδίω την Στεφανή Μπιασόλη, να ευχαριστήσω τους ε, συνεργάτες μας. Ο Τίνο και η Καταρίνα ήταν αυτοί που δούλεψαν σκληρότατα όπως είπες και εσύ. Νομίζω ότι κατά την επεξεργασία αυτού του, ε, αυτής της πρότασης ψηφοφορίας που έχουμε μπροστά μας, καταφέραμε να καταλήξουμε σε καλούς συμβασμούς. Δεν είναι κάτι ε, αυτονόητο. Ε, για την Επιτροπή μας. Διοργανώσαμε δημόσιες ακροάσεις, προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε μια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία προκειμένου να βρεθούν απαντήσεις σε αυτό το, σε αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα το οποίο χαρακτηρίζεται και από διάφορες οπτικές, διάφορα συμφέροντα ε, κάτι το οποίο βεβαίως δεν, δυσκόλεψε, ε, δεν διευκόλυνε το έργο μας για την εξέβρεση συμβιβαστικών λύσεων Γι' αυτό και ενδεχομένως ε, ε, αργήσαμε λίγο. Παρ' όλα αυτά, έγκαιρα πριν από την ψηφοφορία και την απόφαση στο Συμβούλιο, θα καταφέρουμε σήμερα να, ε, καταφέρουμε να, θα καταφέρουμε σήμερα να καταλήξουμε σε μια θετική λύση. οι τροπολογίες βοήθησαν και στην εξισορρόπηση της ε, δικής μας έκθεσης. Υπάρχουν πάντοτε κάποιοι που γελάνε και κάποιοι που κλαίνε. Πάντοτε ε, πρέπει κανείς να είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, ε, ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι 100% ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, είναι η φύση των, ε, των συμβιβασμών αυτή, αλλά νομίζω ότι καταφέραμε να επιτύχουμε μια καλή ισορροπία στο κείμενο αυτό και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν πάρα πάρα πάρα πολύ την, όλη την προηγούμενη χρονιά στο φάκελο αυτό για το σκληρό τους Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Περνάμε στην ψηφοφορία. Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο γρήγορα και όσο πιο προσεκτικά γίνεται. Μπορεί στο ένα ή στο άλλο σημείο να καθυστερήσουμε λίγο, γιατί σε, κάποιες, σε κάποια σημεία ε, θα χρειαστεί να ε, πηδάμε και ορισμένε σελίδες μέχρι να βρούμε την ε, κάθε φορά ε, τροπολογία που θα ψηφίζουμε. Θα προσπαθήσουμε όμως να το κάνουμε γιατί όπως είπα είναι πραγματικά πολύ σπάνιο εδώ στην Επιτροπή Παιδεία και Πολιτισμού να έχουμε μια τέτοια έκθεση μαμούθ, ψηφοφορία μαμούθ. Η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 349 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβασ... Ε, τροπολογία 351 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίστε. Ελπίζω να έχετε τις κάρτες σας. Τοποθετήστε τις, σας παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Α, 378 υπέρ. Κατά. Όχι, συγγνώμη. 378. Επαναλαμβάνω. Τη βρήκατε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 379. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ένβη 20. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 381. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 382 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 383 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 384 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 390 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 391 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 392 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 394 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 397 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 398 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 400. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 401. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, εγκρίνεται. 403 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 405 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 406 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 407 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 408 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική οριζόντια τροπολογία Συμφωνήθηκε αυτό με τους σκιώδεις και περνάμε στην ψηφοφορία. Υπέρ, κατά, αποχές, καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Geschlossen. τη ψηφοφορία. εγκρίνεται με 21 υπέρ 9 κατά. Τροπολογία 409 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Änderungsantrag 65. Τροπολογία 65. 410, Entschuldigung. 410, συγγνώμη. Συγγνώμη, μπερδεύομαι κι εγώ μερικές φορές. 410 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Κανένα πρόβλημα. Ένας ψηφοφορίας. Schlossen. Πέρας ψηφοφορίας. απορρίπτεται με 28 κατά 2 υπέρ. Dann kommen wir zu Kompromiss 8. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Das Ein Kompromiss 8 dafür. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 836. Υπέρ. Ναι, ναι, πρέπει να φιλομετρήσουμε πρώτα εδώ τον πάκο μας. 836. 836.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 Λοιπόν, τροπολογία 837. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 953. Είναι πολύ πιο κάτω στις σελίδες σας.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 Απορρίπτεται. «954 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». «955 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». «956 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». «958 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Γιούρι 55, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήμκο 84, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 957, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήμκο 85, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 960 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουροι. Ψηφίστε παρακαλώ για την, για την τροπολογία 960 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 959 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 961 και Γιούρι 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ήταν πολύ σαφές. Πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 23 23 υπέρ, 7 κατά. Συμβαστική 11. Ψηφίζουμε. Να, τη βρήκα, ωραία. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 964. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14. 13. Όχι, 14. 14. Σωστά το είπα. Α, sind wieder ein paar Seiten dazwischen. Kompromiss 14. Alle gefunden? Συμβαστική 14, τη βρήκατε όλοι. Τέλεια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε στη συμβαστική 16.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 Τι Τη βρήκα. Μου λείπει ένα χαρτάκι. Συμβαστική 16. Κατά, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία. 600 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 425 425. Ξαναλέω. gefunden? Τη βρήκαμε όλοι. Υπέρ. Όχι, να περιμένουμε λίγο ακόμα. Οι σοσιαλιστές δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρούνε την τροπολογία 425. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά.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 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 619 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εντάξει, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσουμε. Geschlossen. Mit 9... Απορρίπτεται. 11 υπέρ, 19 κατά. Περνάμε στην τροπολογία 430. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην τροπολογία 431. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 437 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 438. Α, όχι, όχι. Ε, ταυτιζόταν με την προηγούμενη ακριβώς. Οπότε περνάμε στην 436. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 440. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 457. Δύο σελίδες περίπου παρακάτω. Τη βρήκαμε όλοι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 459 και 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 460 αποσύρθηκε 461 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63. Πρέπει να περάσουμε κάποιες σελίδες μέχρι να βρούμε την τροπολογία 63. Είναι λίγο παρακάτω. Änderungsantrag 63. Alle gefunden? Βρήκαμε όλη την τροπολογία 63. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 566 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 567 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 23, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική 24. Πάλι πρέπει να δείξουμε μερικές σελίδες. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 719. Τη βρήκατε όλοι. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 27. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 749. ...749. Τη βρήκαμε όλοι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 750 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 751 και ΙΜΚΟ 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 757 στην ίδια σελίδα, τουλάχιστον στα δικά μου έγγραφα. Θα ψηφιστούν μαζί με την 763 και η ΙΜΚΟ 76 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 761 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 759 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 764 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 760 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 765 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 762 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 767 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 768 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 769 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 758 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 770 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 771 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 772 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην τροπολογία 786 786. Alle gefunden? 786. Τη βρήκαμε όλοι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήμκο 78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε στην 787 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 793 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 794 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 788 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 789 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 790 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 791 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 792 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 833 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 80. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 8.34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8.35. Και ΙΜΚΟ 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 32. Κομπρομίς 32. Συμβαστική 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική 33. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 35. Περνάμε κάποιες σελίδες και πάλι. Kompromiss 35. Dafür. Συμβαστική 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 1034. Alle gefunden? Τη βρήκαμε όλοι. Ωραία. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1035. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1037. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1036. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1038 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1039 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 1039 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ, 15 κατά, απορρίπτεται. 1040 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, όχι συγγνώμη. Συγγνώμη. Από τη 1040 επειδή εγκρίθηκε περνάμε στην 1043. Μια σελίδα παρακάτω. 1043. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1044. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Συμβαστική 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΜΚΟ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 121. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 41. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 42. Δύο σελίδες παρακάτω, περίπου. Τη βρήκαμε όλοι. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 43. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην ΙΜΚΟ 36. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 300, όχι, λάθος. 143. Περνάμε στην τροπολογία 143. Υπέρ. Τη βρήκαμε όλοι. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λίμπε 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Geschlossen. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 14 υπέρ, 16 κατά. Dann gehen wir zu Liebe 7. Λίμπε 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΕΝΒΙ 9. Ναι, σωστά τα είπα. ΕΝΒΙ 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 150. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γιούρι 7 και 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 9 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 154 και 155 και NV10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12 υπέρ, 18 κατά. 156 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 159. Λίγο παρακάτω. υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 160 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 161 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 162 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. NV12 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 46. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 47. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 177. Λίγο παρακάτω. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 182. Και την 183. Ταυτίζονται. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 185. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Γιούρι 10. Υπέρ. Και 184 μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ένας ψηφοφορίας παρακαλώ ψηφίστε. Geschlossen. Πέρας. Όχι, σαφέστατο ήταν. Συγγνώμη, δεν είδα καλά μάλλον. Θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει αυτό και να είχαμε γλιτώσει το χρόνο. Δεν πειράζει. Ε, 6 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. που ταυτίζεται με την 194. Υπέρ, κατά,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 Συμβαστική 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 222. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία ΙΜΚΟ 21. Λίγες σελίδες παρακάτω. ΙΜΚΟ 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.36 λέει η Πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.37 υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Συμβαστική 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2.43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Κανένα πρόβλημα. Ένα ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ επί της τροπολογίας 2.43. Eine fehlt noch, Κάποιος δεν ψήφισε. Πέρασε ψηφοφορίες. Πέρας, πέρας, πέρας. 22 κατά, 7 υπέρ, απορρίπτεται σαφώς. 244 ή 23 δεν ψηφίζουν. 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 246, 247, ΙΜΚΟ 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 248 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 251 υπέρ. Κατά. 251 ξανά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 249 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 252 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 253 και ΙΜΚΟ 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 254 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 255 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Λίμπε 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήμκο 27 υπέρ. Όχι, συγγνώμη, περνάμε στην συμβαστική 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 12. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Γιούρι 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 264 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 266 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Λίμπε 13 υπέρ κατά αποχές δεν ήταν πολύ σαφές καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ένας της προφορίες ψηφίστε παρακαλώ Geschlossen. Πέρας πληροφορία. 16 υπέρ, 14 κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην 278. 278. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Περνάμε στη 273. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 275. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 280. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 281 περ κατά αποχές απορρίπτεται. 282 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 283 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 284 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.85 και λίμπε 16 υπέρ, 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 298. 298 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, συγγνώμη, απορρίπτεται. απορρίπτεται. 2,99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 16 ταυτιζόταν με την 299, γι' αυτό και περνάμε τώρα στην 303 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 301 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 300 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 17 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορία για την τροπολογία ΛΥΜΠΕ 17. Ψηφίστε παρακαλώ. Ich bin auch schon langsam ein bisschen durcheinander. schließe die Abstimmung. Ja, mit 18 zu 10 abgelehnt. Απορρίπτεται. 10 υπέρ, 18 κατά. Envy 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ωραία, εντάξει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. NV17. Ψηφίστε παρακαλώ. Ένας προφορίας. Πέρας προφορίας. Απορρίπτεται. 10 υπέρ, 19 κατά. Μερικές φορές βλέπω σωστά. Die 304 dafür. 304. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάλι δεν είναι πολύ σαφές. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Geschlossen. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14 υπέρ, 15 κατά. Και περνάμε στην 302 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 305 και λίμπε 18 υπέρ κατά αποχές πάλι δεν ήταν πολύ σαφές καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ Geschlossen. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται 13 υπέρ 16 κατά. Ήμκο 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 306. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 310. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γιούρι 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 311. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 307. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήμικο 31. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λίμπε 20. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Λίμπε 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Γιούρι 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 312 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην ΛΥΜΠΕ 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΛΥΜΠΕ 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.18. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 321 και λίμπε 25 που ταυτίζονται υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 323 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 324 υπέρ, όχι, συγγνώμη, λάθος. Ήμκο 33, ζητώ συγγνώμη, Ήμκο 33 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Λίμπε, όχι, συμβαστική 57, σωστά, στην επόμενη σελίδα, συμβαστική 57, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 338 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 340 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 341 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 342 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 343 και λίμπε 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 344 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 345, 345 υπέρ κατά αποχές 345 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 346 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Λίμπε 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 347 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 348 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε... Αιτιολογικές αναφορές 102 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Λίμπε 1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε στην 96. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 95. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και περνάμε πράγματι στην τελική ψηφοφορία θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ονομαστικά βεβαίω. ναι Die Abstimmung ist geschlossen. Πέραση ψηφοφορίας με 17 υπέρ, 9 κατά και 4 αποχές εγκρίνεται στο σύνολό της η έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε όμως και δεύτερη ψηφοφορία, ονομαστική και πάλι, που είναι για την εντολή για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Κομισιόν βάσει του άρθρου 69 ε, γάμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Ich schließe die Abstimmung. ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 9 κατά, 3 αποχές. Η εντολή ανατίθεται για τις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με διευκολύνατε πάρα πολύ στην ψηφοφορία αυτή. Ήταν πραγματικά ένα δύσκολο έργο, αλλά το επιτελέσαμε όλοι μαζί από κοινού πολύ καλά. Σας διαβεβαιώ, σε σχέση με αυτό που κάναμε μόλις τώρα, η επόμενη ψηφοφορία θα είναι πολύ εύκολη. Σας καθησυχάζω. Να ξαναευχαριστήσουμε άλλη μια φορά την Στεφανή. <laughs> Λοιπόν, έχουμε άλλη μία. Άλλη μία ψηφοφορία. Δεν θα διαρκέσει πολύ ώρα. Ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν από την αίθουσα μπορούν να το κάνουν χωρίς φωνασκίες. Σας παρακαλώ, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Περνάμε στην ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης για την τροποποίηση της οδηγίας 112-216 όσον αφορά τους συντελεστές του ΦΠΑ για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά και μπορούμε να πούμε ότι ο χρόνος βοήθησε να δώσω το λόγο στον ε, ε, εισηγητή, τον κύριο Στρογεύσκη, αν θέλει να πει κάτι. Όχι, δεν θέλει να πει κάτι, οπότε περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 1. Όχι, όχι, όχι, όχι. Περνάμε στην 6. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται. Συγγνώμη. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία, ονομαστική και αυτή. Ένας ψηφοφορία ψηφίστε παρακαλώ. Πέρες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. 30 υπέρ 0 κατά. Θερμά συγχαρητήρια. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, δύο λεπτών, για να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε. Ήταν πραγματικά πολύ κοριστική αυτή η δουλειά που κάναμε. Έχουμε όμως αρκετό χρόνο. Θα συνεχίσουμε σε δύο-τρία λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Und möchte als erstes, äh, einige... Να καλωσορίσω ορισμένους προσκεκλημένους μας. Έχουμε 10 επισκέπτες, φοιτητές από την Γαλλική Σχολή ε, Αγροτικής Ανάπτυξης. Σας καλωσορίζω. Είδατε τις πληροφορίες νομίζω όχι, ε. Ελπίζω, εν πάση περιπτώσει, αυτά που θα συζητήσουμε τώρα ε, να σας κινήσουν το ενδιαφέρον σε έναν βαθμό τουλάχιστον και να αποκομίσετε θετική ε, εικόνα, θετική εντύπωση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας καλωσορίζω. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Γνωμοδότηση πρωτοβουλίας πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξαποστάσεω εκπαίδευση ω μέρος τη Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Διαβίου Μάθηση. Είναι μέρος του πακέτου της οδηγίας για, τα, για τις νέες δεξιότητες. Ε, ο Μίλαν Σβέρ, ο συνάδελφο, είναι ε, συντάκτης της γνωμοδότησης. Θέλω να του δώσω το λόγο απευθείας για να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του. Να σας πω από τώρα ότι η υποβολή για την, ε, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 4η Μαΐου και η ψηφοφορία θα γίνει στις 21 Ιουνίου. Και θα υπάρξει και γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Σβέρ. Παρακαλώ. Äh, äh, äh, ευχαριστώ συνάδελφοι. εκπώνησα ένα σχέδιο έκθεσης ε, για την επαγγελματική κατάρτιση και τη διαβίωματισή ως κομμάτι της ε, γενικότερης στρατηγικής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και το ΕΛΚΙΑ όλες τις προσπαθειές τους και επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες από τη Δημοσιακρόση του Ιανουαρίου έπαιξαν σημαντικό ρόλο για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης, το σχέδιο έκθεσης, το οποίο επίσης περιλαμβάνει τα πρώτα ε, αρχικά σημεία που απαιτούνται για την επιτυχή ανάπτυξη της ε, ε, διαρκούς εκπαίδευσης και της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Αν έχετε σχόλια, αν έχετε οποιασδήποτε βελτιώσεις, τροπολογίες, θα τις δεχθώ ευχαρίστως στην Ευρώπη τα κλασικά πανεπιστημιακά και σχολικά συστήματα έχουν αναβαθμιστεί και μέσω της ε, διαβίου μάθησης. Η διαβίου μάθηση βασίζεται στο γεγονός ότι ζούμε σε μια περίπλοκη ε, κοινωνία υψηλή τεχνολογία, γεμάτη κινδύνους. Γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να μαθαίνουμε διαρκώς, επίσημα, ανεπίσημα, με κάθε ευκαιρία. Όχι μόνο στο χώρο εργασίας, αλλά και στο σπίτι. Δεν πρέπει να πάμε ποτέ να μαθαίνουμε. Είναι σημαντικό για όλους μας. Τα σχολικά συστήματα θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Η πρόσβαση στην ε, εκπαίδευση όταν δεν είναι επαρκής ε, μειώνει, ελαττώνει και το επίπεδο του εργατικού δυναμικού και οδηγεί σε προβλήματα στην οικογένεια και σε κοινωνικό αποκλεισμό. και σε βίαιη ριζοσπαστικοποίηση των νέων, οι οποίοι είναι η πιο ευάλωτη ομάδα. Η πιο εύκολη πρόσβαση στην εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελέσει συνήθη πρακτική και να εγκατασταθεί παντού. Γεγονό που δεν συμβαίνει σήμερα. Γι' αυτό το λόγο η διαβίου μάθηση είναι τόσο σημαντική, διότι παρέχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και βοηθά στη μείωση του κόστους της εκπαίδευσης. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση είναι ο πιο οικονομικός τρόπος σπουδών διότι δεν περιλαμβάνει τις κλασικές δαπάνες των σπουδών. Είμαι βέβαιος ότι οι νέες μορφές διαβίου θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις όπως η υψηλή ανεργία που παραμένει υπερβολικά υψηλή σε μια δεκαετία σχεδόν ε, οι μισές δουλειές που θα υπάρχουν θα είναι, κάτι, θα εντελώς νέες και θα απαιτούν ε, νέα προσόντα. Ε, το πάνω από το 50% των νέων θέσεων εργασίας θα πρέπει να στελεχωθούν από υψηλά καταρτισμένο προσωπικό. Τα πανεπιστήμια πρέπει να εξοπλίσουν τους πτυχιούχους με νέες δεξιότητες και επιχειρηματικές δεξιότητες, ό,τι χρειάζεται για να διεισδύσουν στην αγορά. Στην έκθεση επίσης ε, έχω επισημάνει πόσο σημαντική είναι η εξατομίκευση των σπουδών. Βάσει των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του κάθε σπουδαστή. Αυτή η ευελιξία θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την ποιότητα των σπουδών και να μειώσουμε το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου και των σπουδών στην Ευρώπη, ε, το οποίο παραμένει ακόμα υψηλό. Επίσης πρέπει να πω ότι στην Ευρώπη ελάχιστοι καθηγητές και δάσκαλοι χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία στις τάξεις τους και στα ε, αμφιθέατρά τους, ε, κάτι που πρέπει να υποστηρίξουμε ε, να ενταθεί επίσης ε, ε, η ψηφιακή πλατφόρμα επίσης της τάξης θα αποτελέσει μια γρήγορη απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εποχή της ψηφιοποίησης. Αυτό θα μας βοηθήσει να παρέχουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους και να αντιμετωπίσουμε τους φόβους και τους δισταγμούς. Και σε αυτό εγώ θα, διστασ... θα επικεντρωθώ στην έκθεση. Η έκθεση λοιπόν κάνει έκκληση για την δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαίσιου για όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρχει αραγής λειτουργία της διαβίου μάθησης ε, συμπεριλαμβανομένης ε, της αναγνώρισης των αποτελεσμάτων της άτυπης ε, και της κατά περίπτωση εκπαίδευσης. Πρέπει να διασυνδέονται, πιστεύω, επίσης περισσότερο τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών, ειδικότερα όσον αφορά τις εφαρμοσμένες σπουδές, οι δυνατότητες που παρέχει η εξαποστάσεως εκπαίδευση μέσω του Erasmus Plus θα πρέπει να αξιοποιηθούν και στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει επίσης να προσαρμόζονται στις αλλαγές στην αγορά εργασίας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι και συνεχή εκπαίδευση των διδασκόντων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω σε οποιασδήποτε ε, τροπολογίες και σχόλια. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφοι. Ευχαριστούμε, κύριε ε, Σβέρ. Να δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές για τρία λεπτά ο καθένας. Και ξεκινάμε με τον κύριο Νέκοφ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολύ καλή προσπάθειά του. Σε ό,τι αφορά την μάθηση και την εκπαίδευση εξ και την σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα να πω τα εξής. Η εκπαίδευση εξ είναι ένα εργαλείο χάρη στο οποίο μπορεί να κρατήσουμε τον κόσμο στην ύπεθρο. Επίσης η κατάρτιση εξ αποστάσεως είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση σε μια τέτοια κατάρτιση, ούτω ώστε να μπορέσουν οι νέοι να προσαρμόζονται στις συνεχώς διαφορετικές περιστάσεις καθ' όλη τη διάρκεια του βίου τους. Χρειαζόμαστε τα εξή πράγματα. Καταρχάς εθνικές στρατηγικές, ούτως ώστε να ε, προωθήσουμε τις ψηφιακέ δεξιότητες. Αυτές οι στρατηγικές θα πρέπει να εστιάζουν περισσότερο στο ρόλο του δασκάλου. Ακόμα και στα πλαίσια της ε, μάθησης εξ τα ευρωπαϊκά σχολεία και τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια χρειάζονται καλύτερους δασκάλους, με περισσότερα προσόντα και δεξιότητες, που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Ο κύριος Βέντ πολύ σωστά είπε ότι μόνο το 1 τέταρτο των φοιτητών και μαθητών στην Ευρώπη διδάσκονται από δασκάλους που έχουν πραγματικές ψηφιακέ γνώσεις. Η κατάρτιση των δασκάλων έχει επιδεινωθεί σημαντικά λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ε, γι' αυτό χρειαζόμαστε λοιπόν πόρους όμως για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει να προωθήσουμε μέτρα ούτως ώστε η δουλειά του καθηγητή, η δουλειά του δασκάλου να γίνει πιο ελκυστική. Οι δάσκαλοι σε αεροκατοικημένες περιοχές θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής. Και η εκπαίδευση και η κατάρτιση εξ μπορεί να είναι μια καλή λύση και για αυτούς. Τρίτον, η μάθηση εξ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμπλουτίσει τις γνώσεις και δεξιότητες των ανθρώπων χωρίς να αποβεί αυτό επιζήμιο στην προσωπική τους ισορροπία. Η αγορά εργασίας όλο και πιο πολύ χρειάζεται γνώσεις και δεξιότητες που δεν μπορούν να αποκτηθούν σε μία τάξη. Και ίσως η μάθηση εξ αποστάσεως μπορεί να είναι κατάλληλη. Τέταρτον, αυτά που λέει η έκθεση, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση που θα είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του καθενός και προσαρμοσμένη στις νέες τεχνολογίες, είναι πάρα πολύ σημαντική. Περιμένω να συνεργαστώ πολύ καλά με τον κύριο Σβέν και με τους υπόλοιπους όδης εισηγητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Τζαμάσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Το θέμα αυτής της έκθεσης είναι πολύ σημαντικό. Οι ιδέες του εισηγητή και οι δικές μας προτάσεις θα είναι η κατάλληλη βάση για μια συζήτηση και θα μπορούσαν να δώσουν και κάποια καθοδήγηση, κάποιο προσανατολισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι κοινωνίες μας αλλάζουν συνεχώς. Υπάρχει μια δυναμική αλλαγή και θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Η έκθεση Σβέν είναι πάρα πολύ λεπτομερής και έχει πολύ σημαντικά στοιχεία για το πώς θα αναπτυχθούν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και πώς θα προσαρμοστούν στις ε, τεχνολογικές προκλήσεις. Η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και η ανάγκη για ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών επίσης υπογραμμίζεται στο κείμενο. Συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα online όπου οι εμπειρογνώμονες θα μπορούν εκεί να ανταλλάσσουν τις ε, βέλτιστες αυτές πρακτικές. Για μένα και για την ε, ECR η αρχή της επικουρικότητας όμως είναι πάρα πολύ σημαντική και ελπίζω ότι θα αναφέρεται στην έκθεση στη βέουσα θέση και θα προτείνουμε και τις ε, σχετικές ιδέες στο συνάδελφο. Ε, η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι πρόβλημα σε πολλά κράτη-μέλη. Ε, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε, μπορούμε να προοδεύσουμε χάρη στη συνεργασία. Χρειαζόμαστε μια γενική προσέγγισε ένα πλαίσιο κανονιστικό, μας είπε ο συνάδελφος. Δεν μπορώ να συμφωνήσω όμως με αυτό. Γιατί οι παραδόσεις και η κουλτούρα του κάθε κράτους μέλους είναι τόσο διαφορετικές που ελπίζω ποτέ να μην ρυθμίσουμε τις, ε, τον πολιτισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή τους πολιτισμούς μας. Πάντως θέλω να συνεργαστώ με, με τον συνάδελφο και θα του προτείνω τις ιδέες μας και τις προτάσεις μας. Ευχαριστώ πολύ και περνάμε στον κύριο Κιουτσούκ. Συγγνώμη αν δεν προφέρω σωστά το όνομά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω τον συναδέλφο για το έργο του σε αυτή τη σημαντική έκθεση. Όλε αυτέ οι μορφέ εκπαίδευση μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλά ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, ειδικότερα τα υψηλά επίπεδα τη ενεργεια των νέων σε πολλά κράτη-μέλη, την ασυμφωνία δεξιοτήτων, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου. Εφόσον η εκπαίδευση προσαρμοστεί στις προσωπικές ανάγκες, σε αυτή την ταχύως μεταβαλλόμενη οικονομία, οικονομία αυτές οι νέες μέθοδοι εκπαίδευσης ε, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής, πανευρωπαϊκής στρατηγικής θα μπορέσουν να διευκολύνουν την ε, χωρίς αποκλεισμούς ε, μάθηση για όλους. Ε, συμφωνώ με τον εισηγητή ότι είναι αναγκαία η διαβίου μάθηση στη σημερινή δυναμική τεχνολογικά εξελιγμένη κοινωνία και η εξατομικευμένη αποστάσεως μάθηση προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, κάτι ε, ουσιαστικό, ε, πολύ σημαντικό για ανθρώπους με δικές ανάγκες, ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή που είναι άνεργοι. Έτσι λοιπόν η εξαποστάσεως λοιπον η αποστάσεως μαθηση θα πρέπει να ρυθμίζεται με τους ίδιους κανόνες, όπως και η πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση, αλλά με τα ανάλογα κριτήρια. Θεωρώ ωστόσο ότι περισσότερο εστιάζεται η έκθεση στην εξαποστάσεως μάθηση. Ενώ θα ήθελα εγώ να υπογραμμίζεται εξίσου τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν όσον αφορά την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, την έλλειψη πόρων για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και την ανεπαρκή διαφημισή της και πρόθεσή της είναι αναγκαία η μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και υποστήριξη των φοιτητών μαζί με τη συνεχή αναβάθμιση των διδασκόντων στο πλαίσιο της καινοτομίας και λόγω της ψηφιοποίησης, βαθμιάς ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μαρτίνα Μίχελς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής, κατά τη γνώμη μου, έχει συντάξει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, θέλω να τονίσω ότι φυσικά υπάρχει το δικαίωμα στη διαβίου μάθηση, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μια αντίληψη ότι η διαβίου μάθηση είναι και υποχρέωση. Φυσικά, ε, οι ε, επαγγελματικές απαιτήσει αυξάνονται, ε, αυξάνεται και η ανάγκη για όλο και περισσότερες επαγγελματικές δεξιότητες και την αναβάθμισή τους και την επικαιροποίησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γι' αυτό και πράγματα κράτη-μέλη έχουν ευθύνη να διαμορφώνουν ε, πιο πολύμορφες δυνατότητες ε, μάθησης και εκπαίδευσης. Όπως λέει στο σημείο 4, αυτό ισχύει, αλλά οι αβεβαιότητες δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε, μια, ε, σε έναν ανελαίητο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας, στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει διαρκώς να προσαρμόζονται. Αντίθετα, νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να ε, είναι γνωστές και να διαπιστώνονται τακτικά οι νέες ανάγκες, ιδίως στη διαδικασία και στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης. Πέρα από τις πραγματικά πολύ σημαντικές αλλαγές που θα επιφέρει η ψηφιοποίηση, θα ήταν σημαντικό να υπάρχουν και επιχειρηματικές γνώσεις. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με μια διαδικασία αυτοπροώθησης ε, στην, ε, στην αγορά εργασίας. Νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε και αυτό. Για τις ε, χρηματοδοτικές και διαρθρωτικές προκλήσεις θεωρώ ότι είναι θετικό το ότι η παιδεία ε, χαρακτηρίζεται ως μακροπρόθεσμη επένδυση. Όλες οι μελέτες όμως καταδεικνύουν ότι ό,τι και να κάνουμε στη διαβίου μάθηση δεν πρόκειται να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα αν δεν υπάρξουν επενδύσεις στην προσχολική και στην ε, δημοτική εκπαίδευση. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου πάντοτε τη συνολική εικόνα της παιδείας. Και για το σκοπό αυτό πράγματι είναι χρήσιμη η ευρωπαϊκή ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων και χαιρετίζω τις σχετικές αναφορές του εισηγητή στην, ε, στο σχέδιο έκθεσης του. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Χέλγα Τρούγκε. Ναι, ευχαριστώ για το ζήτημα της, το πολιτικό που αναφέρει και η κυρία Μίχελς. Πιστεύω ότι η διαβίου μάθηση είναι διαρκώς ένα ζήτημα εξισορρόπησης συνδυασμού των, της ανάγκης για απασχόληση. Από την άλλη όμως η διαβίου μάθμιση αφορά την προσωπική εξέλιξη και τη δυνατότητα ε, προσαρμογής στις διάφορες αλλαγές ε, που επέρχονται. Υπάρχει πάντα αυτή η διπλή δομή λοιπόν. Έτσι λοιπόν πολύ γενικά επικροτώ το ότι μα δίνεται αυτή η δυνατότητα να προσφέρουμε περισσότερε δυνατότητε σε ανθρώπου διαφόρων ηλικιών και έχετε δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό φυσικά να ξεκινάμε με τα παιδιά μικρή ηλικία, διότι αυτά αποτελούν ε, τη βάση των πάντων. Δεν πρέπει λοιπόν να τα παραμελούμε σε καμία περίπτωση. Ε, τη... ακούσαμε στις ακροάσεις και οι ακαδημαϊκοί μας είπαν ότι οι ειδικέ δυνατότητες ε, για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και την εξαποστάσεως μάθηση ειδικότερα για νέους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όλες αυτές οι δυνατότητες ε, από την ω μάθηση σε επίσημο πλαίσιο προσφέρει περισσότερες δυνατότητες σε τέτοιους ανθρώπους να αναπτυχθούν, να αναπτύξουν τις ιδέες τους, να επιτυχούν αυτά που επιθυμούν. Τέλος, για μένα ήταν σημαντικό που αντιλήφθηκα ότι για την οικογενειακή ζωή και για τις γυναίκες είναι σημαντικές αυτές οι δυνατότητες εξ αποστάσεως μάθησης διότι έτσι μπορούν να επανασυνδεθούν με τον κόσμο και να βρουν αυτό που επιθυμούν να κάνουν. Επίση, ήταν σαφέ ότι ειδικότερα για του μετανάστε και του πρόσφυγε η εξαποστάσεω μάθηση και οι σχετικέ δυνατότητε είναι κρίσιμη σημασία. Θα επικεντρωθούμε σε αυτέ τι πτυχέ ε, στι τροπολογίε μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλοι δύο μιλητές. Τζούλι Βόρτ και Κριστίνα Λίμπατσκα. Παρακαλώ. Για δύο λεπτά η καθεμία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ έχω δεσμευτεί για τη διαβίου μάθηση. Ε, θεωρώ ότι είναι κρίσιμη σημασία για την σύγχρονη κοινωνία. Αλλά δεν πρέπει να αφορά μόνο τη ε, δουλειά. Αν είναι να σκεφτόμαστε συνεχώ ότι προετοιμάζουμε ανθρώπου να ε, γίνουν ε, κομμάτι ενός μηχαν... μια μεγάλη μηχανή ε, που δημιουργεί όλο και περισσότερο χρήμα, δεν νομίζω ότι πρέπει η διαβίωμα να έχει αυτό το σκοπό. Πρέπει να υποστηρίζουμε τη μάθηση για τη μάθηση αυτή καθεαυτή. Και πρέπει να φροντίσουμε να γίνεται αυτό χωρί αποκλεισμούς, να υπάρχει πρόσβαση για τι γυναίκε, για περιθωριοποιημένες ομάδε και για ανθρώπου μεγαλύτερη ηλικία. Θα ήθελα να σα διηγηθώ μια ιστορία για τον πατέρα μου. Ο πατέρα, μου, ξέρετε, όταν συντοξιδοτήθηκε ως ε, δάσκαλος, ε, έφτιαξε έναν υπολογιστή μόνο του και γνωρίζει περισσότερα για του υπολογιστέ από ότι εγώ. Και όταν τον επισκέφθηκα πριν από λίγου μήνε, είχε εγγραφεί σε ένα online μάθημα για να μάθει πώ να φτιάξει ένα ρομπότ. Και έχει ξεπεράσει τα 80 και δεν το κάνει γιατί θέλει να βρει δουλειά. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι από την κούνια μέχρι το θάνατο είναι πολύ σημαντική η μάθηση ε, και το να προσφέρεται το σχετικό περιβάλλον που ευνοεί κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό. Ε, ήθελα να πω ότι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η έννοια της ε, του επαγγελματικού αλφαβητισμού είναι μια έννοια που μπορεί να εφαρμοστεί άπαντες ανεξαρτήτως φίλου ηλικίας, εθνικότητας, ε, ικανοτήτων. Ουσιαστικά βοηθά να δούμε πώς θα μπορούμε να αξιοποιούμε το χρόνο μας με αξιοπρέπεια και, με, ε, και ποιοτικά ε, και αυτό να ευνοεί την κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ Κριστίνα Λιμπάτσκα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Συνεργάστηκα μαζί του και έχω συνεργαστεί πολλές φορές ε, μαζί του και θεωρώ το σχέδιο εκθεσής του είναι άριστο. Δύο είναι τα θέματα, θεωρώ, που ξεχωρίζουν όσον αφορά την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Δύο πτυχές αυτού του φαινομένου. Έχω ήδη πει σε συναδέλφους ε, σε... πολλές, ε, πολλές φορές ότι ζούμε σε ταχύως μεταβαλλόμενες εποχές ε, το πτυχίο μπορεί να το πάρει κανείς ε, γρηγορότερα από ποτέ. Και λόγω αυτού θεωρώ ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε ορισμένες ε, αξίες, ειδικότερα όσον αφορά τις δεξιότητές μας. Και μετά υπάρχει και η δεύτερη πτυχή που ανέφερε μόλις η Τζούλι η ευκαιρία να κάνει κανείς κάτι για να εξελιχθεί ο ίδιος, κάτι το οποίο παλιότερα δεν ήταν δυνατόν. Η εξαποστάσεω εκπαίδευση παρέχει αυτήν ακριβώ την ευκαιρία να εκπληρώσει κανεί ε, ό,τι τον συναρπάζει. Και συμφωνώ με του συναδέλφου μου που είπαν ότι η υπερβολική νομοθέτηση και ρύθμιση δεν πρόκειται να προωθήσει απαραίτητα περαιτέρω την εξαποστάσεω εκπαίδευση. Ωστόσο, αναμφίβολα πρέπει να παρέχουμε κάποιο κινήτρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι ε, τις σωστές και ε, όρου και απαιτήσει ώστε να αναπτυχθεί αυτού του είδου η εξαποστάσεω εκπαίδευση. Και κάτι άλλο τώρα, η εξαποστάσεω εκπαίδευση είναι κάτι πολύ καλό, διότι διότι περιλαμβάνει εκπαίδευση ε, πολυεπιστημονική ανθρώπους ε, από διάφορους τομείς ε, οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους και επίσης βοηθά τις διάφορες κατευθύνσεις σπουδών και την ανταλλαγή γνώσεων με άλλες χώρες, εμπειριών. Ε, είναι, ιδιαίτερα, είναι πολύ ως μορφή εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν, την κυρία Άντερσον, αν θέλει να λάβει το λόγο για το θέμα αυτό. Είναι ακόμα εδώ μαζί μας. Ωραία, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για το σχέδιο έκθεσης, το οποίο και χαιρετίζουμε ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με το έργο της Κομισιόν στον συγκεκριμένο τομέα. Ευθυγραμμίζεται επίσης και με τις συστάσεις που αναμένουμε να συμπεριλάβουμε στις ανακοινώσεις μας για τον εξοργισμό της παιδείας που θα δημοσιευθεί στις 24 Μαΐου. Να κάνω κάποια συγκεκριμένα σχόλια. Συμφωνούμε απόλυτα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκολυνθεί η διαβίου μάθηση και η κοινωνική ένταξη με την ευρύτατη έννοια. Περιλαμβάνει πρόσφυγες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, όπου βλέπουμε κάποιες ε, πολύ ε, καινοτόμες προσεγγίσεις, αλλά και τους ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Συμφωνούμε επίσης ότι η εξαποστάσεως μάθηση, εκπαίδευση, είναι πολύ σημαντική και συμβάλλει στην ανάπτυξη ε, δεξιοτήτων, στο παγκοσμιοποιημένο υψηλής τεχνολογίας περιβάλλον μας. Επίσης είναι σημαντική η ατομική ανάπτυξη. Δεν, αφορά, δεν αφορά πάντοτε η διαδικασία της μάθησης ε, μόνο και στενά τις ε, επαγγελματικές προοπτικές. Αντιθέτως ε, συμβάλλει και βελτιώνει την προσωπική ικανότητα να ε, αναπτυχθεί κανείς στην κοινωνία, ως μέλος της κοινωνίας. Συμφωνούμε επίσης με την εξατομικευμένη προσέγγιση. Συμφωνούμε επίσης με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, γιατί βλέπουμε πολύ συχνά ε, ότι η καινοτομία πολλές φορές ε, σταματά στα κάμπους των πανεπιστημίων. Χαιρετίζω επίσης την έννοια της διεπιστημονικής γιατί και αυτή είναι πολύ ε, σημαντική, ιδίω για την εξαποστάσεως εκπαίδευση, γιατί χαράσει πολλές φορές και το δρόμο για ε, τα πανεπιστήμια. Άρα θεωρούμε ότι η υψηλής ποιότητας εξαποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει και πρώτη επιλογή, όχι μόνο η απαραίτητα δεύτερη επιλογή, ανάλογα με τις προσωπικές περιστάσεις του ε, κάθε ατόμου. Σε, όσον αφορά τις συστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει μια πρόταση ε, για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας. Ε, εμείς έχουμε μια τέτοια πλατφόρμα η οποία είναι καινοτόμα και η οποία ε, <clears throat> φέρνει μαζί ανθρώπους που εργάζονται στην εκπαίδευση. Ε, σας ευχαριστούμε επίσης για τα καλά σας λόγια για την ε, διαδικτυακή πύλη για τις νέες για τις νέες δεξιότητες. Όσον αφορά την ανταλλαγή πρακτικών, διοργανώσαμε μια σχετική εκδήλωση τον Ιανουάριο που είχε, αφο... που είχε ως θέμα της την ψηφοποίηση στη διδασκαλία και στη μάθηση ε, και το έργο αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Άντερσον. Κυρία Σβέρ, ε, κυρία Σβέρ θέλετε ξανά το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου ξαναδίνετε το λόγο και ευχαριστώ όλους όσοι μίλησαν και συνεργαστήκαν. Είναι ένα θέμα πολύ θετικό, πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο με μεγάλη μου χαρά ανέλαβα το καθήκον του να προετοιμάσω αυτή την έκθεση και διότι μέσω της ε, ε, συνεχούς και εξαποστάσεως εκπαίδευσης μπορούμε πραγματικά να συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για την εκπαίδευση. Η ποιότητα, μια μεγαλύτερη ε, πρόσβαση και στην εκπαίδευση και οι δύο αυτοί τύποι εκπαίδευση μπορούν να μας επιτρέψουν να επιτυχούμε τους στόχους αυτούς. Για να απαντήσω τώρα εν συντομία ε, στα όσα υπόθηκαν εδώ, ελπίζουμε όλοι φυσικά οι νέοι στις γεωργικές περιοχές ε, να παραμείνουν εκεί και οι νέοι συνάδελφοι εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού το υπογράμμισαν. Αλλά για να μείνουν οι νέοι στις αγροτικές περιοχές πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε οι νέοι να ζουν εκεί με αξιοπρέπεια. Ε, να έχουν μια πρόσβαση στην αγορά εργασία. Ε, και ε, το θέμα αυτό είναι διεπιστημονικό. Όταν φεύγουν οι νέοι και σπουδάζουν αλλού αυτό δεν είναι κακό, θα βοηθήσει την μελλοντική τους εξέλιξη. Ε, μιλώντας τώρα για την ψηφιακή πλατφόρμα, ένα, για, ένα γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο, σκοπός μου εδώ δεν ήταν να πω να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εξαποστάσεως εκπαίδευση, για παράδειγμα, καθόλου. Αυτό που ήθελα μάλλον να πω ήταν να δώσουμε ένα κίνητρο στα κράτη-μέλη ώστε αυτά τα ίδια να δημιουργήσουν αυτή τη νομική βάση που απαιτείται. Δεν μιλάμε λοιπόν για εναρμόνιση εδώ, αντιθέτως αυτό που λέμε είναι να έχουμε μια ανάλογη κατάσταση, κατάσταση, κατάσταση από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι κυρίαρχο δικαίωμα, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει κάποιου μηχανισμού που μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη Εδώ μιλάμε λοιπόν για βοήθεια, όχι για παρέμβαση στην εθνική κυριαρχία. Το πλαίσιο αυτό για την εκπαίδευση λοιπόν είναι κάτι επιτυχές. Είναι αδύνατο να φανταστούμε να επιστρέφουν τα πράγματα όπως ήταν πριν. Ε, συμφωνώ με όλους όσοι λένε ότι η αγορά δεν μπορεί να καθορίζει την κατάσταση της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να είναι ο μόνος συντελεστής ε, που θα καθορίζει τις εξελίξεις στην παιδεία. Ωστόσο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αγορά εργασίας διότι η εξέλιξη της οικονομίας ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία ε, και ε, αυτή θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην εκπαίδευση. Φυσικά και δεν είναι ο μόνος που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη, αλλά είναι σημαντικός παράγοντας. Οι πανεπιστημιακοί ε, σπουδαστές ε, δεν αποκτούν μόνο ε, εξειδικευμένες ικανότητες αλλά και γενικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όχι μόνο εκεί που θα εργαστούν αλλά και στην προσωπική του ζωή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για τη συζήτηση. Αναμένω τις τροπολογίες σας και ελπίζω ότι στο τέλος του αυτό το σχέδιο έκθεσης θα ε, καταλήξει να αποτελέσει μια άριστη έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 4η Μαΐου, 2 το μεσημέρι. Εύχομαι σε εσά και τους χειώδεις μια καλή συνεργασία και είμαι βέβαιη ότι θα καταλήξουμε σε μια πολύ θετική έκθεση. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε όλοι σήμερα στις 3 στην κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΚΟΝΤ για, το, για, για να συζητήσουμε το θέμα του Euronews. Συνεδρίαση των συντονιστών θα γίνει στις 11. Γι' αυτό διακόπτεται ε, αυτή τη στιγμή η συνεδρίασή μας και θα συνεχίσουμε στις 11 με τους συντονιστές.